προμοσιευθούν στα πρακτικά της επόμενης Ολομέλειας. Ε, η προθεσμία ε, υποβολής ε, αντίθεσης λίγη αύριο. Επίσης σας λέγω ότι το ΕΛΚ έχει υποβάλει τα ε, ακόλουθα αιτήματα. Ο κύριος Αντώνιο Καντσάν, μέλος της Αντιπροσωπείας για σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο, θα αντικαταστήσει ο κύριο Αλφρέντο Αντωνιώτσι. Ο κύριος Αλφρέντο Αντωνιώτσι ε, θα, θα αντικαταστήσει ο κύριο Καντσάν στην ε, κοινή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Κροατίας. Επίσης, ο κύριος Ανδρέα Κατσολίνα θα γίνει μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών μετά από αίτημα των Σοσιαλιστών. Κύριε Έχετε κάποιο πρόβλημα. Όχι, όχι. Κανεί λοιπόν δεν αντίθεται στις προτάσεις ε, αυτές. Τα πρακτικά της ε, παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν στην έκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου